συνεισφορά θεωρούμε ότι βελτιώνει το κείμενο, από εμάς θα είναι απολύτως αποδεκτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ευχαριστώ τους δύο εισηγητές, τον κύριο Ρωμεύη και την κυρία Ιέρο. Και ευχαριστώ ένθερμα και την Επιτροπή, την εκπρόσωπο από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ σήμερα. Πάντοτε θέλουμε να συνεργασόμαστε μαζί σας. 4 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι, προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Ψηφοφορία στην Επιτροπή 22-23 Ιανουαρίου και προβλέπεται η ψηφοφορία στην Ολομέλεια το Φεβρουάριο. Σα ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 4, πρωτόκολλο μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία τη Γκαμπών. Ε, ε, έχουμε υπογράψει 24 Απριλίου το σχέδιο του πρωτοκόλου και το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ προσωρινά. Ο κύριος στόχος του πρωτοκόλου είναι να δοθούν ε, αλευτικές δυνατότητες σε 35 σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ύδατα της Γκαμπών σύμφωνα με τις καλύτερες δυνατές επιστημονικές συμβουλές και συστάσεις του ICAT. Κατόπιν της παρουσίας της Κομισιόν και την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε στις 3 Οκτωβρίου, Σήμερα τον κύριο Φεραίρα θα, εκπροσωπήσει η κυρία Ζούμπερ. Και έχω την τιμή να της δώσω το λόγο. Ευχαριστώ. Αντικαθιστώ τον κύριο φερείρα και θα ήθελα να σας ε, διαβιβάσω τις κύριες ανησυχίες του σε σχέση με αυτή την ελληνική συμφωνία. Όπως σας είπα αυτή η νέα συμφωνία εγκρίθηκε στις 24 Ιουλίου, θα διαρκέσει τρία χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας. Η νέα συμφωνία προβλέπει ελευτικές δυνατότητες για τις ακόλουθες συμφωνίες. 27 ψυγεία και 8 σκάφη ε, που αλλιεύουν με καλάβι. Δεν έχει ανανεωθεί η δυνατότητα για τα παραγαδιάρικα και η αντιπαροχή που θα καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1.350.000 ευρώ και αυτό το ποσό έχει εγκρίνει 20.000 τόνους αναφοράς που ανταποκρίνεται σε στο ποσό των 900.000 ευρώ σε σχέση με την πρόσβαση στους ελευτικούς ε, πόρους. Επίσης υπάρχει υποστήριξη για την των μερικής ελευθερικής πολιτικής της Γαμπών ε, μέχρι 350.000 ευρώ. Ο εισηγητής ε, συστήνει την έγκριση αυτού του πρωτοκόλου και κάνει και κάποιες σκέψεις τις οποίες θα σας αναφέρω. Αφενός θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η προώθηση η Καμπον να ερευνήσει τους ίδιους ε, πόρους της ε, και για την κατανάλωση αλλά και για την εξαγωγή. Ο εισηγητής θεωρεί ότι οι κανόνες εκφόρτωσης δεν σέβονται τους στόχους αυτούς και προτείνει να δημιουργηθούν συνθήκες που θα επιραίνουν την, να καταστούν επιχειρησιακά οι δομές στους λιμένες και να γίνεται η εκφόρτωση ε, πληρώνοντας τέλη στην Καμπόν. Επίσης θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να Υπάρχει παρακολούθηση ε, των σκαφών που αλεύουν στα ύδατα της Γκαμπών. Θεωρεί ότι είναι απαραίτητη τη διαφάνεια της διαδικασίας και του προσδιορισμού των συνολικών ελευμάτων. Αυτή η διαφάνεια πρέπει να βελτιωθεί καθώς και τα μέτρα καταπολέμησης ε, της ε, αλίας Αγιουγιού. Και τέλος, ο συγητής πιστεύει ότι θα πρέπει να, ληφθεί υπόψη, να ληφθούν υπόψη πλήρως τα σημεία 2 και 3 ε, του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται πλήρως για όλα τα στάδια των διαδικασιών που σχετίζονται με το πρωτόκολλο ή με την ανανέωσή του. Προτείνει στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο ετήσια να παρουσιάζεται μία έκθεση για το πολιετές ε, σχέδιο που αναφέρεται στο άρθρο 7 του πρωτόπουλου όπως και να υποβάλλεται και η δήλωση αλλιευμάτων. Να γίνεται σεβαστή υποχρέωση αυτή η υποβολή στις δήλωσης αλλιευμάτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και... Η κυρία Φράγκα έχει καταρχήν το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Ζούμπερ που αντικαταστήσε τον κύριο Φερέιρα. Ο κύριος Φερέιρα αναφέρεται στο πρόβλημα των υποδομών στην Καμπόν. Δεν ε, υπάρχουν λιμάνια στην Καμπόν όπου μπορούν πραγματικά να εκφορτώνονται τα αλλιεύματα του κοινοτικού στόλου και Γι' αυτό μέχρι τώρα έχει χρησιμοποιηθεί το λιμάνι της Αμπιτζάν στην ακτή του Αλαφαντοστού. Όπως και να έχει το πρωτόκολλο προτείνει, καθώς δεν μπορεί να, να επιβάλλει υποχρεώσεις εκφόρτωσης, γιατί είναι αδύνατη η εκφόρτωση, αλλά λέγεται στο κείμενο ότι στην περίπτωση που οι λιμενικές υποδομές είναι επιχειρησιακές, τότε υπάρχει υποχρέωση εκφόρτωσης. Δηλαδή, από τη στιγμή που λειτουργούν οι υποδομές αυτές, έχουμε αυτή την υποχρέωση εκφόρτωσης από τον κοινοτικό στόλο. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα στην Καμπόν, ότι οι 12 ε, βιομηχανίες που υπήρχαν έχουν οικονομικά και διαφορετικά προβλήματα πάρα πολύ σοβαρά και επομένως έχουν σταματήσει τις εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2010. Είχαμε και πτώχευση της ε, μεγαλύτερης εταιρείας. Στην Καμπόν όμως ε, υπήρξε δυνατότητα στο παρελθόν εξαγωγή, Το πρόβλημα είναι ότι πτώχευσαν οι επιχειρήσεις. Όμως εμένα αυτό που με ανησυχεί είναι η εφαρμογή αυτού του κανονισμού σε σχέση με την παράνομη λαθρέα και άναρχη ελίας. Από όσο γνωρίζω εγώ δεν έχει τεθεί ακόμα σε εφαρμογή ε, το σύστημα των πιστοποιητικών της πιστοποίησης των ελευμάτων. Πότε προβλέπετε λοιπόν κάτι τέτοιο μπορεί να μας ενημερώσει η Κομισιόν. Όπως ε, είπαμε, αυτή η συμφωνία αφορά τον τόνο, ιδιαίτερα μεταναστευτικά είδη, ρυθμίζεται από τον ΆΙΚΑ τη συμφωνία αυτή και τα είδη αυτά και δεν θέτει κάποιο πρόβλημα ε, γιατί ε, δεν υπάρχει εμπλοκή με την αιρεσιτεχνική αλία στην Καμπόν. Εγώ ελπίζω να βελτιώσει τελικά η Γκαμπών τις υποδομές της, έτσι ώστε και ο κοινοτικό στόλος να μπορεί να προβαίνει σε εκφόρτωση στην Γκαμπών, για να μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε και την μεταπητική βιομηχανία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πάντως εγώ συμφωνώ με το πρωτόκολλο και υποστηρίζω όσα λέει ο εισηγητής. Να υποστηρίξουμε δηλαδή αυτό το πρωτόκολλο αλίας. Ευχαριστώ κυρία Φράγκα, κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ. θα ήθελα να επανειληφθώ. Να σας πω ότι υποστηρίζω αυτή τη συμφωνία, η οποία είναι σημαντική για τα θηναλιευτικά του Ευρωπαϊκού Στόλου. Και θα ήθελα να τονίσω ότι ο προϋπολογισμός και τα κονδύλια θα αυξήσουν τη συνεισφορά των ε, εφοπλιστών. Ε, υπάρχει δέσμευση τουλάχιστον από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Στόλου προκειμένου μαζί με τις αρχές και τους υπεύθυνους να βελτιωθεί η αηφορία και η ενημέρωση. Ε, υπάρχει και κάτι που δεν νομίζω δεν αναφέρθηκε για τις 450.000 ευρώ για ε, την υποδομή των λιμένων και ακούσαμε ότι δεν είναι επαρκή η ανάπτυξη αυτού του τομέα στην Καμπόν. Να τονίσω επίση ότι αυτό το πρωτόκολλο, το πρωτόκολλο δηλώνει μία δέσμευση για την πρόθεση μιας υπεύθυνης αλίας ε, με σεβασμό στις συστάσεις του ICAT και η εκπόνηση ενός πολιετούς τομεακού προγράμματος θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη το στρατηγικό σχέδιο για την Καμπόν. Και όλα αυτά και φυσικά ενισχύοντας και τη συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να εξαλειφθούν και τα προβλήματα της παράνομης αλίας. Νομίζω ότι βέβαια δεν ξεκινούν αυτά τα προβλήματα από τα ευρωπαϊκά σκάφη. Επομένω, υποστηρίζουμε την έκθεση αυτή και συμφωνούμε με τον εισηγητή. Thank you, Chair. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την αντικαταστάτρια ε, της κυρίας Φεραίρα για την παρουσίαση. Συμφωνώ απόλυτα με τις ε, ανησυχίες που εξέφρασε η κυρία Φράγκα και τις ε, στηρίζω σχετικά με την εκφόρτωση και την έλλειψη υποδομών στην Καμπόν. όσον αφορά τους λιμένες και πιστεύω πως θα ήταν καλό η τομεακή στήριξη στη συμφωνία αυτή να στοχεύει στην βελτίωση της ε, υποδομής των λιμένων. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή εάν όντω ισχύει αυτό, εάν υπάρχει κάποια σχετική συζήτηση με την Καμπόν για αυτό. Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει κατά πόσο η νέα αυτή συμφωνία, το νέο αυτό πρωτόκολλο, θα συντονίζεται με το ενδέκατο πρόγραμμα χρηματοδότησης EDF και εάν θα υπάρχει συνεργασία και συντονισμός με τις ε, πολιτικές ανάπτυξης και συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείτε, θα ήθελα να μάθω το βαθμό με τον οποίο συντονίζουμε τις ενέργειες αυτές. Επίσης, ε, η γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού τονίζει ότι όλα τα αλληλευτικά σκάφη που υπάρχονται στο πρωτόκολλο πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσει ε, υποβολής αναφοράς. Θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή αν υπήρξαν κάποια προβλήματα με αυτές τις ε, αναφορές στο παρελθόν. Επίσης, η κυρία Φερέιρα ανέφερε ένα μεγάλο ποσοστό παραλιεύματος ε, καρχαριών. και καρχαρία ως αλλιευόμενο είδος. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλληλεία καρχαρία σύμφωνα με την συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ιζαμπέλ Τομά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον εισηγητή και την εκπρόσωπό του σήμερα να ξεκινήσω εκφράζοντας τη λύπη μου για το γεγονός ότι παλιμπεδίζει το κοινοβούλιο σε αυτή τη στιγμή. Και το λέω γιατί η Κομισιόν μας είχε στον αέρα τα τελευταία δύο χρόνια με μερικές ψηλοπληροφορίες που μας είδαινε έτσι ώστε να μην μπορούμε εμείς να παρακολουθήσουμε τις διαπραγματεύσεις σαν να είμαστε μικρά παιδιά και πιστεύω πως καλό είναι να μας τηρείτε πιο ενήμερους για να γνωρίζουμε τι πρόοδο σημειώνουν αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και ένα δεύτερο για να συμφωνήσω με την Ισαμπέλ και για την Αλία Καρχαρία. Ξέρετε τι γίνεται για το πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα παραγάρια σε καρχαρίες και ε, θα ήθελα να μου πείτε και οι τράτες αυτές επίσης ε, τι τύχεις θα τύχουν. Θέλουμε μια βελτίωση της ε, συμφωνίας. Ξέρετε πως είχαμε την ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα οποία είχαμε κρατήσει στον αέρα τη συμφωνία την υποχρέωση εκφόρτωσης τη συζητήσαμε. Παρ' όλα αυτά χρειαζόμαστε περισσότερες προφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άκουσα τι είπαν οι συνάδελφοι για τον φάκελο, για την αναπτυξιακή βοήθεια και το κατά πόσο θα χρηματοδοτήσει υποδομές. Το 20% επίσης που ακούστηκε ως ποσό μας ικανοποίησε. Επίσης το μητρό, το ηλεκτρονικό μητρό αλίας, ε, το οποίο αποτελεί ε, ως υποχρεωτικό ημορολόγιο μία βελτίωση. Ε, όλα τα σχετικά με, τις, με τα πληρώματα των σκαφών επίσης μας ικανοποιούν η έλεγχη και η βελτίωση αυτών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, Όλα είναι σημαντικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Και θα ήθελα να συγχαρώ τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο την Κομισιόν. Το πρωτόκολλο λοιπόν όπως διαπραγματεύτηκε και η έκθεση να ξέρετε ότι από μένα θα στηριχθεί. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι λοιπόν έλαβαν το λόγο για το θέμα, για τη συμφωνία με την Καπών. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όλα τα ερωτήματα που έχουν γίνει. Θέλω να ευχαριστήσω όμως καταρχήν και την Επιτροπή Ανάπτυξης και ε, Προϋπολογισμού και εσάς βεβαίως ε, για μια έκθεση η οποία είναι θετική. Για τις ερωτήσεις που μου κάνατε, το πρωτόκαλο αυτό αναφέρεται με συγχωρείτε, δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο, συγκεκριμένη διάταξη για την εκφόρτωση, μια και δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι λιμένες. Δηλαδή, θα συμπεριλάβουν την υποχρέωση αυτή όταν χτιστούν τα λιμάνια και οι υποδομές τους. Και να σας πω πως από την πλευρά της Γκαμπών ανέλαβαν να προχωρήσουν μέσα στα επόμενα τρία χρόνια με την διαμόρφωση των λιμενικών ε, υποδομών έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες αλίας. Αυτό λοιπόν θα οδηγεί σε μια προσαρμογή ε, της ε, του βασικού εμπορικού λιμένα της χώρας προς αυτή την κατεύθυνση. Η παράνομη, η λαθρέα αλία είναι ένα πρόβλημα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως οι αρχές της χώρας αυτή τη στιγμή έχουν αποκτήσει όλα τα εργαλεία έτσι ώστε να δημιουργήσουν την αρμόδια αρχή η οποία θα παραδίδει αυτά τα πιστοποιητικά έτσι ώστε να καλύπτουμε τις υποχρεώσεις μας ώστε να καταπολεμήσουμε τη λαθρέα και άνερχη αλληλεία. Η Γκαμπόν αποφάσισε να στηρίξει κυρίως δύο κλάδους. Πρώτα απ' όλα τον έλεγχο των αλληλευτικών δραστηριοτήτων και δεύτερον την βελτίωση των, ε, της παρακολούθησης έτσι ώστε να αυξηθούν οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Λορίν ρώτησε πώς μπορούμε να ε, συνεργαστούμε με το Ταμείο. Πρέπει να σας πω πως εδώ για την Καμπόν δεν πρόκειται για χώρο προτεραιότητας. Εμείς θέλουμε να τα δούμε τα θέματα περιφερειακά περισσότερο και νομίζω ότι αυτό ζήτησε και ο εισηγητής. Σας ενημέρωσε πως υπάρχει και ένα συγκεκριμένο άτομο βέβαια αρμόδιο για τη διαχείριση αυτής της συμφωνίας. Βρίσκεται στη Λιμπρεβίλ και αυτό θα μας ε, διευκολύνει στο να ε, συντονιστούμε καλύτερα με, τη διεθνή, με το Διεθνή Οργανισμό. Τώρα, είπατε πως ε, υπάρχει ένα είδος παλιμπεδισμός ή ότι σας μεταχειριζόμαστε σαν να είσαστε παιδιά. Νομίζω ότι ότι αυτή η σιγεία σειρμάτου έχει να κάνει με το ότι η Γκαμπόν δεν ερχόταν να διαπραγματευτεί. Και γι' αυτό δεν σας είχαμε πει τίποτα. Τώρα, για το ηλεκτρονικό ημερολόγιο πλοίου, για το Μητρό αυτό, στη Μικτή Επιτροπή που συναντήθηκε 28 και 29 Οκτωβρίου, σας στείλαμε καταρχήν τα πρακτικά και για το θέμα αυτό θα εγκατασταθεί για το 2014. Έχουμε συμφωνήσει το χρονοδιάγραμμα με τις αρχές της χώρας και αυτή τη στιγμή κάνουμε την προσευχή μας όλα να λειτουργήσουν. Είμαι στη διάθεσή σας, σας ευχαριστώ. Euh, ευχαριστώ, Κριστιαν. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ζούμπερ αν θέλει να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ. Όχι, θέλω απλώς να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Ε, θα τα διαβάσω στον κύριο Φερέιρα. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε κυρία Ζούπερ που αντικαταστήσατε το συνάδελφο. Να περάσουμε τώρα στην έκθεση Λοβίν ε, για την υγεία των Και ότι αυτή η γνωμοδότηση είχε ανατεθεί Στου Πρασίνου, στι 4 ε, Οκτωβρίου είχαμε κάνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και νομίζω ότι η κυρία Λοβίνα μπορεί να μα παρουσιάσει σήμερα την γνωμοδότησή τη. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε πρώτα την Ιζαμπέλ και κατόπιν του υπόλοιπου συναδέλφου. Συγγνώμη. 2 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία κατάσταση τροπολογιών για την έκθεση Φερέιρα. Ιστορική ημερομηνία για τη Γαλλία για τον Αστερίξ. Για τη μάχη του Άστερλιτς, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Καταρχήν. Να σας πω ότι καλωσορίζω αυτή την πρόταση για ένα νέο κανονισμό για την υγεία των ζώων που θα πλουστεύσει την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τον έλεγχο και την πρόληψη των οσων και θα καταργήσει πάνω από 40 οδηγίες και πολλές εκατοντάδες κατεξουσιοδότηση πράξεις και όλα αυτά θα συγκεντρωθούν σε ένα κανονισμό. Όμως ε, η πρόκληση απλούστευσης είναι ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι καλύπτονται όλα τα στοιχεία των διαφορών θετημάτων και ότι παραμένει συνεκτικό το κείμενο και παραμένει και ευέλικτος ο νέος κανονισμός και ικανός να καταπολεμήσει αναδυόμενες ε, νόσους και απειλές για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων. Στην έκθεσή μου Ίσως ε, να σας φανεί ότι υπάρχουν πολλές τροπολογίες, αλλά βασικά καλύπτουν ε, τρία θέματα και υπάρχει και μια κάποια επαναληπτικότητα, καλό, καθώς ε, οι ίδιοι όροι έχουν ελαχθεί σε διάφορες παραγράφους. Το πρώτο θέμα αφορά τη σύνδεση μεταξύ της υγείας των ζώων και της προστασίας, της ε, καλής μεταχείρισης των ζώων, αν θέλετε. Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση της Κομισιόν. Θα είναι το νομικό πλαίσιο για να υποστηριχθεί η στρατηγική για την υγεία των ζώων που δημοσιεύτηκε το 2007. Όμως το πεδίο εφαρμογής περιορίζεται στις μολυσματικές νόσους. Όλοι μας όμως γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας ε, ισχυρός συνδέσμος μεταξύ της υγείας των ζώων και της προστασίας των ζώων της ευημερίας των ζώων. Αν υπάρχουν ζώα που υποφέρουν ή βιώνουν πολύ μεγάλο άγχος, φυσικά είναι πολύ πιο ευάλωτα σε νόσους. Ακόμη και αν γνωρίζουμε λοιπόν ότι η Κομισιόν σκοπεύει να προτείνει ένα νέο κανονισμό σε σχέση με την προστασία, την ευημερία των ζώων, πρόταση από τον καλωσορισμό, πιστεύω ότι ένα σύνδεσμο μεταξύ τη υγεία και τη προστασία των ζώων πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στον κανονισμό αυτό. Επομένω, έχω κάνει αναφορέ στην τροπολογία 1, σε μια θεολογική σκέψη τη Συνδίκης τη Λισαβόνας, όπου το άρθρο 13 δηλώνει ότι σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων. Και νομίζω ότι στους στόχους της πρότασης θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η βελτιωμένη για τον ζώων είναι ένας από τους στόχους, όχι μόνο η καλύτερη ανθρώπινη υγεία ή το να βελτιώσουμε την οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μία προσθήκη λοιπόν σε μία τροπολογία. Και κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικός ο στόχος αυτός. Ε, Αν έχουμε ένα κανονισμό για την υγεία των ζώων θα πρέπει αυτό να συμπεριλαμβάνεται και μεταξύ των στόχων. Και ε, στις τροπολογίες 9 ε, ως 11 έχουμε ακριβώς την ίδια ανησυχία για την υγεία και την προστασία των ζώων. Το επόμενο θέμα είναι το θέμα των αντιβιωτικών η Παγκόσμιο Οργάνωση Υγείας ε, λέει ότι η διάδοση της ανθεκτικότητας στα αντιβιωτικά είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές κατά της ανθρωπότητας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από 25.000 άνθρωποι ετησίως ε, καταλήγουν λόγω από μολυσματικέ νόσου που προκαλούνται από βακτηρία που έχουν ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά και ε, τα αντιβιωτικά που χρησιμοποιούνται στα ζώα ε, που χρησιμοποιούνται για παραγωγή τροφίμων ευνοούν τη διάδοση των βακτηρίων στην τροφική αλυσίδα. Επομένω, είναι πολύ σημαντικό και για τα ζώα, αλλά και για την ανθρώπινη υγεία, και για τη ζωική και για την ανθρώπινη υγεία να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τη χρήση των αντιβιωτικών από την υδατοκαλλιέργεια γνωρίζουμε ότι βελτιωμένη η διαχείριση και όταν ε, έχουμε μικρότερες πυκνότητες ηχθείων και, και εισαγωγή εμβολίων μπορεί αυτό να οδηγήσει σε μειωμένη χρήση των αντιβιωτικών. Στην ακρόαση ε, που έλαβε χώρα πριν δύο μερές στην Επιτροπή Γεωργίας, ένας από τους εμπειρογνώμονες ε, έδωσε παράδειγμα πώ η χρήση των αντιβιωτικών στην παραγωγή σολομού στην Νορβηγία οδήγησε σε μείωση από 40 τόνους αντιβιωτικά φτάσανε στη χρήση 40 κιλών ε, αντιβιωτικών. Έχουμε δηλαδή μείωση 99%. Και καθώς αυξήθηκε η παραγωγή από 20.000 τόνους ε, ψάρια της ΙΟΥ σε 1 εκατομμύριο έτσι λοιπόν βλέπουμε τεράστια βελτίωση στη μείωση της χρήσης αντιβιωτικών. Και είδα και αυτό το ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση για την ε, ε, χθιοκαλλιέργεια στη Φιλανδία. Εκεί η χρήση των αντιβιωτικών ήταν πολύ ψηλή. Εκεί υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης. Πιστεύω λοιπόν ότι η υπεύθυνη χρήση των αντιβιωτικών θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη στον κανονισμό αυτό. Επίσης αυτό πιστεύει και ο συγητή από την Επιτροπή Γεωργίας. Διευρύνοντας λοιπόν τα μέτρα για να καλύψουμε και τη χρήση των κτηνιατρικών προϊόντων σε όλες τις ε, μεταδοτικές νόσους ε, και όχι μόνο αυτές το παράρτημα, θα αντιμετωπιστεί η χρήση των αντιβιωτικών. Και αυτή είναι η λογική που διέπει τις τροπολογίες μου για τα άρθρα 46 και 47. Τώρα, τελευταία θεματική αφορά το πεδίο εφαρμογή. Στην πρόταση της Κομισιόν θεωρώ ότι οι ορισμοί προκαλούν σύγχυση και δεν είναι ξεκάθαρο πότε ο κανονισμός καλύπτει τους ηχθείς και τα στρακόδερα για τα ενιδρία ή τα ζώα που κρατώνται, που εχμαλωτίζονται από τον άνθρωπο πριν ε, τη σφαγή ή πριν την απελευθέρωση στη φύση. Για μένα είναι σημαντικό ότι ε, όσοι ε, κρατούν ψάρια, πέρα από αυτούς που ασχολούνται με την κολλιέργεια και αυτοί έχουν ευθύνες Επίσης, ε, οι νόσοι προκύπτουν και από ψάρια που μπορεί να βρίσκονται σε νηδρία ή στα σπίτια ή στα εστιατόρια και ξέρουμε ότι σε ορισμένε περιπτώσει αναπελευθερώνονται στη φύση από αλείς ε, ή από αριστέχνες αλείς ε, που προσπαθούν να εισαγάγουν νέα είδη μπορεί να προκαλούνται νόση. Έτσι λοιπόν έχω διαγράψει ένα τμήμα του ορισμού στο άρθρο 4.5 της πρόταση της Κομισιόν όπου ορίζονται ε, τα υδρόβια ζώα μόνο αυτά που είναι ζώα υδατοκαλλιέργειας. Και έχουμε και το ίδιο να συμβαίνει στα ορισμό για τα kept animals, τα ζώα που είναι υπό εχμαλωσία. Οι τροπολογίε μου που αφορά τα άρθρα που ρυθμίζουν τις ε, μετακινήσεις ε, των ζώων μεταξύ κρατών μελών, άρθρα 1, 196 ε, μέχρι 200 έχει ως στόχο να προστατεύσει τους πληθυσμούς άγριων ζώων από τις νόσους. Εγώ θεωρώ ότι θα ήταν σαφέστερος ο κανονισμός αν χρησιμοποιηθεί η ορολογία processing establishment όπως έχουμε και στην οδηγία για το 2006 καθώς ε, η σφαγή ε, των ε, ζώων αυτών γίνεται σε τέτοιες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και όχι σε εγκαταστάσεις που ορίζει αυτός ο κανονισμός για να καταλάβουμε καλύτερα τις απαιτήσει και τις ευθύνε όσων σφαγιάζουν ζώα η εγκαταστάση, μάλλον θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο όρος της εγκατάστασης μεταποίησης μαζί με τον όρο aquatic food establishments, δηλαδή εγκαταστάσεις ε, για τα ε, υδροβια ζώα. Αυτά από μένα και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν να λάβουν το λόγο. Δεν βλέπω κάποιον. Θα δώσω το, το λόγο λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν σας έχω ξεχάσει, μην ανησυχείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την συγγήτρια για το έργο της για την προετοιμασία αυτού του σχέδιου έκθεσης. Βεβαίω, είμαστε ικανοποιημένοι που η συγγήτρια βρήκε μόνο τρία καυτά σημεία στην πρόταση της Κομισιόν. Η πρόταση της Κομισιόν είναι πάρα πολύ φιλόδοξη, όπως είπα και η ίδια η συγγήτρια. Γι' αυτό είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που υπάρχει από την πλευρά της ε, υποστήριξη στη γενική συλλογιστική της πρότασης ε, και υπάρχουν μόνο κάποιες ανησυχίες σε σχέση με το πρόβλημα σχέση μεταξύ της υγείας των ζώων και της προστασίας ή ευημερία των ζώων. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα καυτό θέμα. Εμείς ε, πιστεύουμε ότι το έχουμε ξεκαθαρίσει αρκετά καλά. Αυτή είναι μια πρόταση που αφορά την υγεία των ζώων και ιδίως την καταπολέμηση των μολυσματικών νόσων. Φυσικά, ορισμένες πτυχές της σχέσης μεταξύ υγείας και καταπολέμησης των μολυσματικών νόσων και της Προστασία των ζώων, τη ευημερία των ζώων υπάρχουν, όμως πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να αφήσουμε στη μελλοντική πρόταση της Κομισιόν για την προστασία των ζώων τη ρύθμιση των ε, σημαντικών πτυχών σε σχέση με το θέμα αυτό. Διαφορετικά, εδώ κινδυνεύουμε να ανοίξουμε μία συζήτηση που θα είναι πολύ πιο δύσκολη δεδομένης της ευαισθησίας της προβληματικής της προστασίας των ζώων. Έχοντας και κατά νου ποια είναι αφενός τα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να δούμε σε σχέση με την προστασία των ζώων, αλλά αφετέρου και ποια είναι τα όρια που η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει σε σχέση με τη δυνατότητα ανάληψης δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της προστασίας των ζώων. Σε ό,τι αφορά τώρα το πρόβλημα της εφεκτικότητας στα αντιβιωτικά. Είναι πολύ πολύπλοκο το πρόβλημα αυτό και θέλω να τονίσω την ανακοίνωση της Κομισιόν που δημοσιεύτηκε πριν δύο χρόνια σε σχέση με την ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά. Εκεί απαριθμούσαμε μία σειρά δράσεων ε, σε σχέση με την αυθεντικότητα στη βιωτικά, 12 δράσεις αν θυμάμαι καλά και μόνο μία από αυτές αφορά το σχέδιο κανονισμού που έχουμε ενωπιών μας σήμερα. Ακριβώς γιατί η Κομισιόν σκοπεύει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό της ε, ανθεκτικότητας αντιβιωτικά σε πολλά μέτωπα. Το καινοτόμο στοιχείο στην πρόταση της Κομισιόν είναι μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των κτηνιάτρων, των κτηνοτρόφων, όλων όσων ε, ασχολούνται και με την υδατοκαλλιέργεια για να υπάρχει μια σωστή χρήση των αντιβιωτικών σε ό,τι αφορά τώρα τις νόσους που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο και εδώ μπαίνουμε σε κάτι πολύ σημαντικό. Ίσως θα μπορούσε να είναι και κάπως ε, αμφίσιμο το θέμα και αναφέρουμε σε κάποιες τροπολογίες που προτείνει η συγκεκριά, θα μπορούσε να είναι κάπως αμφίσιμο, τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν κάπως να μπερδευτούν αν επιβληθούν μέτρα σε σχέση με τη χρήση των αντιβιωτικών και για όσους που δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο, γιατί είναι ενδιαφέρον την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα, να θέσει προβλήματα. Όμως, ε, σε γενικές γραμμές, ε, θέλουμε να συζητήσουμε περαιτέρω με την εισηγήτρια τις ιδέες που έχει προτείνει σε σχέση με μια πιο ορθή, μια πιο σωστή χρήση των αντιβιατικών. Είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα αυτό, το τονίζω και η Κομισιόν προσδίδει τη μέγιστη σημασία. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή και του ορισμού, Πιθανότατα η συγκήτρια έχει δίκιο. Ίσως ε, κάτι πρέπει να προσαρμόσουμε σε σχέση με την έννοια το ποια υδρόβια ζώα πρέπει να θεωρηθούν ότι είναι υπό τον έλεγχο του ανθρώπου. Η λύση που έχετε προτείνει μας προβληματίζει κάπως. Θα θέλαμε να τη συζητήσουμε περαιτέρω με την εισηγήτρια για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη διατύπωση του κειμένου σε ό,τι φορά τώρα τις εγκαταστάσεις. Ευχαριστώ να σας δώσουμε εξηγήσει. Πιστεύουμε ότι ο ορισμός που προτείνεται από την Κομισιόν είναι ο σωστός. Όμως θα θέλαμε να το συζητήσουμε περαιτέρω με την εισηγήτρια. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Merci Σας ευχαριστώ πολύ. Ισαμπέλ, έχεις κάτι να προσθέσεις. Απλώς να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχόλια που έκανε. Εξακολουθώ να πιστεύω πως υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να αναφερθούμε στην ευζοία των ζώων ως ένα από τους βασικούς λόγους που προκαλούν ασθένειες στα ζώα, γιατί αν δεν διαβιώνουν σε καλές συνθήκες τότε η υγεία τους κινδυνεύει αλλά καταλαβαίνω ότι στους στόχους αυτό θεωρείται και κουτί της πανδώρας, το οποίο ενδεχομένω δεν θέλετε να ανοίξουμε. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει πως η ανθεκτικότητα στα μικρόβια αποτελεί πια μεγάλο πρόβλημα και πως στον κανονισμό αυτό θα καταφέρουμε να το αντιμετωπίσουμε. Για το πεδίο εφαρμογή και τους ορισμούς Ας συνεργαστούμε. Ευχαριστώ. Ωραία. Σας υπενθυμίζω πως προθεσμία για τις τροπολογίες έχουμε το μεσημέρι της 4ης Δεκεμβρίου, 4 Δεκεμβρίου λοιπόν, 12 το μεσημέρι. Για να κλείσουμε λοιπόν το πρωινό, έχουμε την έκθεση για την αντιπροσωπεία που πήγε στην Δανία 28 με 30 Οκτωβρίου πήγανε στην Βόρεια Γιουτλάνδη τρεις συνάδελφοι πήγαν από εδώ η οποία συντονίστηκε από, την συνάδελφο, από τον συνάδελφο Όλη Κρίστανσεν στον οποίο θα ήθελα να μεταφέρετε τα συγχαρητήριά μας και νομίζω ότι αν διαβάσετε τα πρακτικά θα ενημερωθείτε για το τι συνέβη. Ήταν πραγματικά πολύτιμη η συμβολή αυτής της αντιπροσωπίας και θεωρώ πως ήταν πάρα πολύ πετυχημένη. Ο Γκαμπριέλ Μάτ, ο αγαπημένος πρόεδρος, παρόλο που δεν ήταν εκεί και δεν είναι και σήμερα εδώ, μου ζήτησε να χαιρετήσω τα αποτελέσματα και γι' αυτό και εγώ με τη σειρά μου θα σας συγχαρώ. Εάν θέλετε, κάποιος από την αντιπροσωπεία μπορεί να πάρει το λόγο για να μας εξηγήσει τι συνέβη σε αυτό το τόσο ενδιαφέρον ταξίδι. Δεν ξέρω με ποιον θα ξεκινήσουμε, με τις κυρίες, μια και σήμερα έχουμε ξεκινήσει με τα γυναικεία θέματα. Ντολόρες, θες να ξεκινήσει, συμφωνία ο συνάδελφος. Μα όταν είναι δύο gentlemen δίπλα μου, πώς μπορώ να πω όχι. Μου ζήτησαν να δώσω κάποιες πληροφορίες ε, από τη γραμματεία γιατί ο κύριος Ολέ λείπει. Τι να προσθέσω. Αυτά που είπατε κι εσείς. Δύο μέρες πήγαμε με ένα πρόγραμμα εξαιρετικά σφιχτό. Και πιστεύω πως πραγματικά οι υπηρεσίες ε, της Επιτροπής ε, εργάστηκαν καταπληκτικά για να τα καταφέρουμε με αποτελέσματα πολύ θετικά. Πήγαμε στο Τεχνολογικό Ίδρυμα για την Αλληλεία, πήγαμε στην Ένωση Αλλιέων, πήγαμε και επισκεφτήκαμε διάφορα έργα ε, με συνεταιρισμούς σε μικρά μέρη, όπου μία γυναίκα που ήταν η καπετάνισσα μας εξήγησε τι έκανε με τις μικροπιστώσεις που έλαβε που έφτιαξε κάποια σκάφη μεταποίησης γιατί μιλάμε για παράκτια αλληλεία και τα εμπορεύεται και στην τοπική αγορά τις ανάγκες που είχαν για στήριξη αυτά τα μέρη, γιατί κατά παράδοση ζουν από την αλληλευτική βιομηχανία και από την αλληλεία και νομίζω ότι η επίσκεψη αυτή μας γέμισε ικανοποίηση. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσω και τον δόκτωρα Κριστίμερμαν για το πώς έχει η Βαλτική, πώς είναι σήμερα η Βόρειος Θάλασσα. Έχουμε δει φωτογραφίες και από τις δικές μας θα διαπιστώσετε πως η εμπειρία αυτή ήταν πραγματικά πολύτιμη. Είδα πως τελικά η ανησυχία των μικρομεσαίων αλλιέων είναι πάντα η ίδια, όπου και να βρίσκονται. Πως δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν πόρους. Και χρειάζεται ίσως εμείς να ευαισθητοποιηθούμε περισσότερο εμείς γιατί έχουν λιγότερα μέσα για να οργανωθούν, δεν μπορούν να μας πιέσουν σε εισαγωγικά τόσο εύκολα. Δηλαδή βρίσκουν τρόπους για να επιβιώσουν και μας λέγανε πως οι νέοι δεν θεωρούν την αλληλεία ελκυστική γιατί είναι τόσο δύσκολες οι συνθήκες οπότε μας ζήτησαν και εκεί να τους βοηθήσουμε. Από αυτό λοιπόν ορμόμενοι μία ακόμα έκκληση ευαισθητοποιηθείτε γιατί είναι ένα πρόβλημα που έχουμε παντού. Επαναλαμβάνω και πάλι πως δίνω τα συγχαρητήριά μου στον κύριο Ολέ που το οργάνωσε, στην Επιτροπή και σε όλα τα άτομα που εργάστηκαν και που μας βοήθησαν που παρόλο το φοβερό κρύο του Βορρό, γιατί καταλαβαίνετε πόσο κρύα έκανε, να τα καταφέρουμε σε τόσο λίγο διάστημα να κάνουμε τόσα πολλά πράγματα. Ευχαριστώ, Ντολόρες. Θέλεις και εσύ το λόγο, Άντωνη. Ναι, ευχαριστώ και εγώ θα συνταχθώ με τα όσα είπε η Ντολόρες Γκαρσία Ιέρο. Η αντιπροσωπεία αυτή, κατά τη γνώμη μου, κάλυψε όλους τους στόχους της. Το πρόγραμμα ήταν αρκετά ποικιλόμορφο και ήταν πολύ αποτελεσματική η οργάνωση που έγινε και κυρίως από τον Όλη Κρίστενσεν. Πήγαμε και στο λευτικό Πάρκο της Βόρειας Θάλασσας. Εκεί έχουμε ένα ίδρυμα, ένα φορέα που ασχολείται με την καινοτομία στην Αλία και με την έρευνα. Συνδυασμός ε, δημόσιας και ιδιωτικής πρωτοβουλίας που μας έδειξε τι κάνει, πώς λειτουργεί. Είδαμε πώς λειτουργεί μια δεξαμενή σκέψη, ένα think tank. γιατί έχουν ένα τμήμα που κοιτάνε εργαλεία λίας, ε, τεχνολογία κτλ. έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερο επιλεκτικά. Πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία αυτή. Και είχαμε και την ευκαιρία να συναντηθούμε με την συμβουλευτική υπηρεσία του ΙΣΕ, με τον Οργανισμό για την Αλληλεία στη Βόρεια Θάλασσα, που ακούσαμε με πολλές λεπτομέρειες το τι συμβαίνει με το γάδο και τη βιωσιμότητα των αλευτικών πόρων. Πολύ χρήσιμα. Πολλά από τα σχόλια που έκαναν για τη βιολογική εξέλιξη του είδους και για το πώς λειτουργεί το ICA ήταν ε, σημαντικά. Είδαμε και τους εκπροσώπους του φορέα ε, που ε, κάνει την θυσία για την βιολογική αλληλεία που έχει δύο ετικέτες, μία για την βιώσιμη αλληλεία και μία για τη βιολογική. Τους ρωτήσαμε τι γίνεται με την αλληλεία μικρής κλίμακας, εάν είναι πολύ βαρύ για τους μικρούς αυτούς επιχειρηματίες να ζητήσουν να πιστοποιηθούν, εάν αξίζει. Επίσης είδαμε το θέμα της εκφόρτωσης και αν αυτή η ε, οικολογική, βιολογική με συγχωρείτε ετικέτα χρησιμοποιείται. Επίσης τους μιλήσαμε για την μεταρρύθμιση που κάνουμε εδώ. Ήρθαμε σε επαφή με εκπροσώπους του κλάδου να μας πούν τα βιώματά τους, τις ποσοστώσεις λοιπά Αν στην Δανία έχουν δει όλα αυτά να φέρνουν μια συγκέντρωση της αλληλείας, πήγαμε σε μια καινοτόμα εγκατάσταση για ηχθειοκαλλιέργεια σολομού που βρίσκεται στη φάση της ε, εγκατάστασης και γίνεται σε κλειστές εγκαταστάσεις. Αυτή είναι η διαφορά. Και μας εξήγησαν τι κάνουν με ευρωπαϊκή στήριξη και πήγαμε και σε κάποιες εγκαταστάσεις που έχουν θαλάσσιες δραστηριότητες. Πήγαμε και είδαμε το ωκεανιάριο που βοηθάει αυτές τις ε, θαλάσσιες, για να τις χαρακτηρίσω έτσι, οι θαλασσοπόρες κοινότητες, με πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα. Βλέπεις τι κάνει μια μικρή κοινότητα με ένα μικρό λιμάνι, δηλαδή βγάζαν, βγάζαν τραβούσαν τις βάρκες στην άμμο και ξεφόρτωναν έτσι, ένας περίεργος τρόπος. Πώς εμπορεύονται κατευθείαν τα νοπά προϊόντα πώς προσθέτουν νοπά, πώς, με πώς ε, εμπορεύονται τα προϊόντα τους, πώς τα προωθούν. Όπου η αλληλεία δεν είναι μόνο για την επιβίωση οικονομικός πόρος, αλλά τρόπο ζωής. Για μας που είμαστε από το νου το, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς λειτουργεί η αλία στο βορρά. Σε χώρες όπως η Δανία. Όπου γύρω από την αλία έχουμε μία σειρά φορείς, οργανώσεις, πρωτοβουλίες, ιδιωτικές και δημόσιες, οι οποίες προσπαθούν να συνδέσουν αυτή την οικονομική δραστηριότητα με το σύνολο της κοινωνικής ζωής. Μία επίσκεψη λοιπόν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, πολύ θετική και για τους ομολόγους μας, γιατί τους εξηγήσαμε πού έχουμε προχωρήσει, πού πάει η μεταρρύθμιση, ποια θέματα είναι υποσυζήτηση, ποιες είναι οι διάφορες απόψεις. Να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις που αισθάνονται για να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια, περισσότερη ευκρίνεια και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Οι ίδιοι σε όσα κάνουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ Αντολίν για την παρέμβασή σου και ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, για όλες τις ε, παρεμβάσεις τους που μας παρουσίασαν αυτή την ενδιαφέρουσα αποστολή στην Ενία. Τώρα πρόκειται ε, για το επόμενο θέμα. Είναι μια άλλη αποστολή που αφορά το ICAT, μια αποστολή όπου συμμετείχαν η Κάρμεν Φράγκα, ο Γκαμπριελ Μάτο και ο Ραουλ Ρομέβα στο Cape Town, στην Νότια Αφρική, την περασμένη εβδομάδα. Θα τους δώσω το λόγο, ξεκινήσω με την κυρία Φράγκα για να μας πει ποια είναι τα αποτελέσματα. Και φυσικά και ο Ραούλ θα πάρει το λόγο, ο Γκαμπριελ Έχουμε κάπως διαφορετικές απόψεις, επομένω ε, καλό θα είναι να πάρουμε και δύο το λόγο. Ευχαριστώ καταρχήν τον κύριο Μπελαρτινέλη, ο οποίος συνέταξε ένα σημείωμα που έχει διαναμηθεί σε όλους, έτσι λοιπόν δεν αναφερθώ σε όλα τα σημεία, αλλά θα επικεντρωθώ στα πιο ενδιαφέροντα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις και τα λοιπά. Η Κομισιόν δεν είναι εδώ, μπορώ να σκίσω κριτική χωρίς κανένα πρόβλημα. Καταρχήν, Πρέπει να σας πω ότι για του χρόνου, για τα περισσότερα από θέματα, υπήρξε ένα rollover, μία μετακίνηση, γιατί θα υπάρξει μία αξιολόγηση για τα αποθέματα, για τα περισσότερα αποθέματα φέτος. Επομένως, οι αποφάσεις θα ληφθούν του χρόνου. Αυτό να το ξέρετε ότι η συνεδρίαση του ICAT ε, θα είναι πιο ενδιαφέρουσα του χρόνου από ότι φέτος. Ε, θα αναλυθούν διάφορα είδη, ο ερυθρός τόνος, ε, ε, της Ανατολής, της Δύσης κτλ. Όμως ε, θέλω να αφαιρθώ στον ε, ερυθρό τόνο. Υπάρχει ένα σχέδιο αποκατάστασης, θα αξιολογηθεί ο ερυθρός τόνος ε, του χρόνου, όμως φέτος υπήρχε μια πρόταση της Ιαπωνίας όπου προτινόταν αύξηση 400.000 τόνους, Δηλαδή από 3.300 περίπου 3.800. Κατά τα λοιπά δεν υπήρχαν μεγάλες τροποποιήσεις στην πρόταση. Τώρα οι περισσότεροι ήταν υπέρ αυτής της μικρής συμβολικής ε, αύξησης ε, γιατί δεν θεωρούταν ότι θα μπορούσε να υπάρχει ε, κάποιο πρόβλημα. Επομένως, ουσιαστικά ήταν κάπως σε μια ειδοποίηση. Είπαμε ότι είμαστε σε μια ε, εποχή αλλαγής και μπορεί να δοθεί μια ελπίδα στον τομέα. εγώ είμαι πιο ριζοσπαστική από τον κύριο Ρωμέβα, όμως υπόθηκε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα από το σχέδιο αν του είχαν δοθεί και 100 γραμμάρια, ούτε τότε θα είχαν δεχτεί, γιατί εδώ δεν υπάρχει ευελιξία. Έτσι λοιπόν, από την στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε όχι, όχι, όχι, όχι. Επομένως, ε, πέρα από ότι όλοι ε, ε, ήθελαν μια τάση αύξησης, υπήρχε αυτή η διαφοροποίηση. Υπήρχε βέβαια και ένα δεύτερο σημαντικό θέμα, μια πρόταση του Καναδά, για την τροποποίηση της περίοδου απαγόρευσης αλίας στις ζώνες όπου για βιολογικούς λόγους και όπου έχουμε ιδιαίτερα μεταναστευτικά ήδη δεν μπορεί να γίνει αλίευση του ερυθρού τόνου ακόμη και αν υπάρχει ποσόστοση κτλ. Αυτό συνέπτε με έτοιμα από τις ε, περιφερειακές οργανώσεις που επίσης έχουν το ίδιο πρόβλημα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντί να είναι λίγο πιο ευέλικτη όταν επιπρόσθετα οι Ηνωμένε Πολιτείε και θυμάμαι πολύ καλά ήταν υπέρ της πρότασης του Καναδά και είχε πει ότι όταν δεν μιλάμε για ζώνες αναπαραγωγής θα υπήρχε μια ευελιξία στο άνοιγμα των απαγορευμένων περιοχών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλεγε όχι, όχι, εγώ δεν θέλω αλλαγές. Και τελικά αυτό οδήγησε στο εξή αποτέλεσμα. Ο Καναδάς ε, τελικά εξανάγκασε να γίνει μια ψηφοφορία που την κέρδισε κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό ήταν κάπως περίεργο, ε, γιατί ο Καναδάς επέμενε να γίνει η ψηφοφορία και τελικά κέρδισε με συντριπτική πλειοψηφία και πραγματικά η Κομισιόν έμεινε σε μια γελία θέση γιατί δεν υπεράσπισε συμφέροντα που είχε παρόμοια με της Νορβηγίας αφενός από την άλλη δεν είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το πρόβλημα αυτό και τελικά την τελευταία μέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου τα κράτη-μέλη να μην επιτεθούν στον κύριο Ντεπίπερ, κατέθεσε μια τροποποίηση που μπήκε στο σχέδιο αποκατάστασης έτσι ώστε περιοχές όπως η Ασόρες ή τα Κανάρια να μπορούν να ζητήσουν από την Κομισιόν ε, να κάνει κάποιες μικρές τροποποίησεις. Αυτά για να σας δώσω μια ιδέα για το πώς γίνεται η διαπραγμάτευση και καθώς εμείς είμαστε παρατηρητές εκεί και εγώ εδώ έχω την υποχρέωση να κάνω κριτική σε αυτές τις διαπραγματεύσεις που δεν θεωρώ ότι ήταν και θεαματικές. Τώρα, το θέμα των 300 ε, τόνων δεν έγινε δεκτό γιατί το απέσυρε η Ιαπωνία. Και το Μαρόκο έκανε μία ερώτηση στην Επιστημονική Επιτροπή, η οποία είπε ότι αυτή 400 τόνοι θα σήμαινε μία διαφοροποίηση των 2,9% και ήταν εντός του ορίου που μπορούσε να γίνει αποδεκτό που είναι 5% για να μην υπάρχουν μεγάλες αλλαγέ. Δηλαδή η Τεχνική και Επιστημονική Επιτροπή δεν είχε κανένα πρόβλημα να το δεχθεί αυτό, αλλά νομίζω ότι μπροστά στην άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ιαπωνία αποφάσισε να το αποσύρει και να περιμένει το επόμενο έτος. Οπότε και φαίνεται ότι οι δυνατότητες αύξησης θα είναι μεγαλύτερες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ε, τηλεσκοπικές κάμερες, ε, αρέσει πολύ στον κύριο Ρωμέβα αυτό το θέμα, καλύτερα να σας το εξηγήσει ο ίδιος. εμάς. Ε, μας ενδιαφέρει από ελευτικές άποψεις, λοιπόν ο ερυθρός τόνος ε, των δυτικών υδάτων. Και επίσης η διαχείριση των καρχαριών είναι ένα θέμα που μας συναρπάζει. Εδώ εμείς ε, ήμασταν αντίθετοι σε μια πρόταση της Κομισιόν για τα πτερίγια, όμως ζητήσαμε τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το ίδιο πάθος που υπεράσπιζε εδώ την πρότασή της να την υπερασπίζει και στα διεθνή φόρα. Δυστυχώς όμως δεν το είδαμε αυτό γιατί πάντοτε σχεδόν πηγαίνει εκεί, low profile και μας λέει ότι δεν θέλω καν να μιλήσω για αυτό το θέμα. Παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Ένωση τρει προτάσει Η μία ήταν επέκταση τη Ευρωπαϊκή ε, Πολιτική ε, για τα πτερίγια. Ούτε καν πέντε λεπτά δεν άντεξε γιατί βγήκαν η Ιαπωνία και άλλοι με τα ίδια επιχειρήματα που έχουμε αναφέρει και εδώ και ένα από αυτό το επιχείρημα όταν καν πήγε στην ομάδα εργασία. Και κατόπιν άλλα δύο θέματα που τα παρουσιάζουν ενίοτε, που είναι να περιοριστεί το επίπεδο ε, της ε, αλίας τελικά ε, η θέση του Καναδά και των ασιατικών χωρών για ένα συγκεκριμένο είδος, την υποστηρίζει όμως για τη λάμνα. Με συγχωρείτε, με παίρνουν τηλέφωνο, λέει ο μιλήτρια. Ούτε αυτό το επιχείρημα πέρασε. Τώρα, επίσης, μένει το θέμα του ελέγχου. Είναι και αυτό ένα θέμα με την Κάνα που μας ε, ντροπιάζει γιατί ξέρετε ότι την Κάνα ποτέ δεν σέβεται τα μέτρα του ICAT και μάλιστα εδώ και καιρό. Ε, ε, Επομένως, προφανώς τέθηκε το ζήτημα της Γκάνας και πρώτη φορά υπήρχε εκεί και ο Υπουργό τη Γκάνας γιατί ενδιαφερόταν πάρα πολύ να επελυθεί το θέμα αυτό. Όπω ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χάρη σε κάποιε καταγγελίε τη Ισπανία, διερευνά το ζήτημα αυτό και χάρη στον κανονισμό της παράνομης λαφρέας και άνομης, παράνομης ερευνά τι μπορεί να κάνει με την Γκάνα. Η Γκάνα εκεί είπε ότι είχε μία ικανότητα που δεν αναφέρεται στο Μητρό, ότι είχε 13 σκάφη ενώ υπάρχουν 17 στο Μητρό και κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εμείς είχαμε εγκαταστήσει ένα σύστημα παρακολούθηση σκαφών που δεν λειτουργούσε. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είπε ότι τίποτα δεν είχε εγκαταστήσει. Λοιπόν, ε, τώρα για να συνοψίσω, για να καταλάβετε εκεί, ε, το κύριο ζήτημα είναι ε, η κάρτα ταυτοποίησης, δηλαδή φτάνουμε στο τελευταίο στάδιο πριν από την απαγόρευση εξαγωγών και υπάρχει πάντοτε μία σειρά χωρών που υποστηρίζουν την Κάνα για διάφορα εμπορικά συμφέροντα και για άλλα παρόμοια συμφέροντα και τελικά απλώς αυτό που έγινε ήταν ότι έγινε μία προειδοποίηση. Αυτά όμως συμβαίνουν και εγώ ήθελα να τονίσω αυτά τα σημεία και θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο για τι διατάξει αλίας και για άλλα θέματα. Θα τα αφήσω να τα σχολιάσει ο κύριο Ρωμέβα που του αρέσουν και πολύ και θα τα πει καλύτερα από μένα. Όπως είπατε λοιπόν πολύ σωστά Κάρμεν, ακούσαμε εσά και μετά το συνάδελφο. Κάρμεν, δεν είναι ποτέ σχεδόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ευέλικτη, οπότε με το που το επιβεβαιώσατε. Επίσης, ε, επιβεβαιώθηκε η Προεδρία για δύο χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, Ραούλ, το λόγο. Αυτά τα οποία διηγήθηκε η Κάρμεν είναι αλήθεια. Εγώ απλώς έχω την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δύο προβλήματα. Καταρχήν ο ερυθρός τόνος που είναι ε, το πιο σημαντικό από αυτά, το εμβληματικό είδος και για το σχέδιο για την περιοχή που μας ενδιαφέρει είπαν δεν θα μετακινηθούν. Αυτό είναι, αυτό είπαν τα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και εκεί θα παραμείνουμε. Τώρα, για τη συγκεκριμένη σύσταση της Επιστημονικής Επιτροπής, εκεί ήταν να μην έχουμε καμία αύξηση ποσόστοσης φέτος. Αυτό έλεγε απερίφραστα η Επιστημονική Επιτροπή. Δεν ήταν δηλαδή έλλειψη ευελιξίας, γιατί είπε πως ενώ έχουμε σημάδια πως το απόθεμα περνάει σε μια ενδεχόμενη ε, αναγέννηση, φάση αναγέννησης, πως παρόλα αυτά χρειαζόμαστε συνέχεια στην ε, υιοθέτηση των μέτρων, άρα λοιπόν δεν προτείνει την αύξηση των ποσοστώσεων. Το είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά κυρίως η Επιστημονική Επιτροπή. Είχαμε βέβαια στην Ιαπωνία που έλεγε 400 τόνους παραπάνω γιατί έχουμε μελέτες που μας το επιτρέπουν και υπήρχαν και άλλες χώρες όπως η Τουρκία, η Λιβύη, η Αλγερία, το Μαρόκο που έλεγαν αφού έχουμε ανακτήσει τα αποθέματα ας δρέψουμε το πλεονέκτημα, ας αυξήσουμε τις ποσοστώσεις και δεν λέγανε 400 τόνους, λέγανε πολύ παραπάνω. Εάν λοιπόν αυξήσεις 400 εκατομμύρια, επειδή το μεγαλύτερο τμήμα ανήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έμενε πολύ λίγο για τους υπόλοιπους. Το οποίο, εάν δεν είχαμε μια πραγματικά μεγάλη ε, αύξηση του ΤΑΚ, δεν θα κάναμε τίποτα αληθεύει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πολύ λίγο χώρο ευελιξίας. Πρώτον για τα όσα είπε η Επιστημονική Επιτροπή και δεύτερον για τα όσα ζητούσαν τα άλλα κράτη. Τελικά συμφωνήθηκε το 2014 να γίνει μια ενημέρωση στα πλαίσια του τρέχοντος σχεδίου και το 2015 μια αξιολόγηση αποθεμάτων για να δούμε πώς πηγαίνουν έτσι ώστε από αυτή την επανεξιολόγηση να ορίσουμε τα καινούρια τάκ και τις καινούριες ποσοστώσεις. Άρα λοιπόν η επόμενη χρονιά για τον ερθρό τόνο από θέματα της Ανατολής είναι πολύ σημαντικό γιατί θα προχωρήσουμε επαναλαμβάνω σε επανεξιολόγηση αυτών. Για τον ερυθρό τόνο του Ατλαντικού που επίσης είναι σημαντικό το θέμα των στερεοκοπικών ε, Καμερών, που είναι ένα πρόβλημα. Γιατί θέλουμε να γνωρίσουμε πόσα, πόσα ψάρια και τι ψάρια μπαίνουν, ας πούμε, στις παγίδες. Πόσα περνάνε από τα δίχτυα. Γιατί ο τρόπος υπολογισμού σήμερα είναι φοβερά ανακριβής. Οι διαστάσεις που μας δίνουν δεν είναι αξιόπιστες. Άρα λοιπόν, τελικά, το περιθώριο λάθος είναι πολλά πολυτόνι. Πρότεινε λοιπόν να χρησιμοποιεί αυτή την στερεοσκοπική κάμερα κάποιο σκάφος που επιτρέπει να υπολογίζει καλύτερα τους τόνους που περνάνε πριν ξεκινήσει η πάχυνση ε, στις παγίδες, στα κλωβιά. Οπότε, στο σχέδιο για την ανάκαμψη των αποθεμάτων Για την περιοχή των Αζόρων είχαμε ένα σημείο σχετικό και η πρότασή μου είναι αφού θα χρειαστεί να προσαρμόσουμε την πρόταση αυτή του ICAT και που λόγω ε, προβλημάτων χρόνου δεν μπόρεσα να προετοιμάσω σήμερα για να ε, ψηφιστεί εδώ, να το καταθέσουμε ως προφορική τροπολογία να ψηφιστεί για την Ολομέλεια έτσι ώστε να κατασταλάξουμε σε ένα συμβιβασμό που θα μας επιτρέψει την πρόταση αυτή για τις στερεοκοπικές κάμερες να την εντάξουμε. Γιατί είναι ένα τεχνικό θέμα που μπορεί να μας ε, λύσει κάποια προβλήματα. Ένα θετικό λοιπόν για τη συζήτηση που έγινε για την Ορβηγία και αυτή είναι μια προσωπική άποψη, το γεγονός πως η χώρα αυτή παραδοσιακά αισθάνεται ότι την έχουν κακομεταχειριστεί ε, οι υπόλοιποι, δεν ξέρω αν αυτό εσείς το ε, συμμερίζετε, πρέπει να αναγνωρίσουμε πως προσπάθησε να μας πιέσει, ε, τα στήλωσε και κέρδισε. Για τον τόνο, τον δυτικό τόνο, Κάποια από τα συμβαλόμενα μέρη θέλουν εκεί να αυξηθούν τα αποθέματα και θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Έχουμε ξεκινήσει να έχουμε αρκετά αξιόπιστα στοιχεία πως τα δύο αποθέματα αυτά, ανατολικά και δυτικά, είναι πιο συνδεδεμένα από ό,τι πιστεύαμε. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν εάν τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα ανάλογα με την περιοχή του τόνου γιατί βλέπουμε πως τουλάχιστον ένα κομμάτι του πληθυσμού όχι αυτή η οποία ζει στη Μεσόγειο, αλλά μία η οποία είναι νομαδική, η οποία μεν περνάει από τη Μεσόγειο, αλλά φεύγει κατευθείαν ε, προς τις δυτικές περιοχές και αυτό χρήζει αξιολόγηση. Αυτά για τον ερθρό τόνο. Πού ήταν το πιο εμβληματικό στοιχείο. Τώρα για τους καρχαρίες, ναι, είναι λυπηρό που μετά από πέντε χρόνια συγκεκριμένων προτάσεων δεν κάναμε τίποτα. Νομίζω πως αυτό είναι ένα μεγάλο σφάλμα και θα πρέπει να αξιολογήσουμε το αν έχουμε ακολουθήσει την κατάλληλη πορεία. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υπερασπίστηκε το θέμα με το πτερίγιο. Η δική μας θέση είναι πολύ σκληρή σε σχέση με αυτή που έχουν ο Καναδάς και οι ασιατικές χώρες. Τώρα για τον Ξηφία, εδώ έχω ένα στοιχείο που μου φαίνεται σημαντικό. Εάν για τον ερθρό τόνο λέμε πως η Επιστημονική Επιτροπή υποβάλλει συστάσεις και λέει αυτά τα τάκ και ποσοστώσεις δεν θα πρέπει να ε, αλλάξουν, υπάρχει, υπάρχουν κάποιες χώρες που θέλουν να ευελι να γίνει πιο ελαστική η οριοθέτηση των ποσοστώσεων και νομίζω ότι για τον Ξηφία, αυτό έγινε για τους τόνους, έγινε σχεδόν το αντίθετο. Δηλαδή, η Επιστημονική Επιτροπή είπε πως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, κάποιες περιστάσεις επί τις οποίες ε, πάνε καλύτερα από ό,τι είχε υπολογιστεί και ήταν όχι ο ίδιος ο κλάδος αλίας που είπε όχι, πρέπει να είμαστε πιο συνετοί και να εφαρμόσουμε ποσοστώσεις περιοριστικές γιατί τα πράγματα με τον ξηφία δεν είναι και τόσο ρόδινα. Ένα συγκεκριμένο μέτρο επίσης είναι το θέμα της προστασίας της χελώνας, της θαλάσσιας χελώνας που εμάς δεν μας αφορά ιδιαίτερα. Άλλα συμβαλόμενα μέτρα ε, μέλη, ναι, αλλά είπαμε ότι θα μπορούσαμε ε, την παρεπίπτουσα αλληλεία χελώνας να τη μειώσουμε. Εκεί πρέπει να δούμε τι γίνεται με τον έλεγχο. Το πρόβλημα που έχει ο ICAT, γιατί δεν ξέρω τις άλλες οργανώσεις, το μεγάλο πρόβλημα του ICAT είναι πως αντί να γίνει μία εξασφάλιση ότι δεν έχουμε λαθραλία ή άναρχη αλληλεία. Έχει καταλήξει ένας οργανισμός που όλα αυτά τα κρύβουμε κάτω από το τραπέζι. Και μου το είπε προσωπικά κάποιος και δεν θα τον κατονομάσω, είναι ότι κάποιος μου είπε ότι πέρσι μόλις έμαθε πώς λειτουργεί αυτό. Όταν μια χώρα παραπονέθηκε πως έλαβε κάρτα προειδοποίησης. Είναι, η Σενεγάλη ήταν αυτή. Και παρόλο που κάποιοι ε, πιστεύουν ότι προσπαθεί, ε, είπε η Σενεγάλη σας παρακαλώ στηρίξε με. Και κάποιοι την στήριξαν. Όταν λοιπόν αυτό το συμβαλόμενο μέρος παρουσίασε αυτές τις επιστολές στήριξης, στηρίχθηκε και από όσους είχε η ίδια χώρα στηρίξει στο παρελθόν. Τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, το ένα χέρι είναι το και τα δύο το πρόσωπο. Το πρόβλημα είναι το σύστημα. Είναι ένα σύστημα όπου τελικά δεν έχουμε εργαλεία αρκετά ισχυρά για όσους ε, ανεύθυνα αντιμετωπίζουν το θέμα της λαθρέας αλληλείας και της άναρχης αλληλείας. Το πρόβλημα για μένα είναι ο έλεγχος. Ο ICAT δεν είναι ένας χώρος αρκετά αξιόπιστος έτσι ώστε να καταπολεμήσει τέτοιου είδους αλία. Η Γκάνα δεν είναι τυχαία περίπτωση. Έχουμε αυτό το, αυτή την εβδομάδα, λάβαμε τον κατάλογο, τον τελικό κατάλογο που, των χωρών που θα αντιμετωπίσουν κυρώσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδεχομένως. Και είναι όντως η Γκάνα. Και επειδή ήταν πραγματικά επιθετική σε όλες τις διαπραγματεύσεις η Γκάνα, Πιστεύω πως η πρόθεσή της ως χώρα ήταν σαφής. Να καταφέρει εκεί να στηρίξουν την Κάνα οι υπόλοιπες αφρικανικές χώρες και να παραστήσει πως είναι η φωνή της Αφρικής. Δηλαδή να έχουμε μία ε, περιφερειοποίηση μέσα στις περιφερειακές οργανώσεις αλίας. Δηλαδή να μην εκφράζει μόνο την Κάνα αλλά και τις άλλες αφρικανικές χώρες. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα που για μένα είναι το πιο σημαντικό για τα επόμενα χρόνια. Με λίγα λόγια λοιπόν, η συνεδρίαση ήταν η συνηθισμένη. Είναι η τελευταία που πήγα ως Ευρωβουλευτής και νομίζω ότι ακολουθήσαμε τη γνωστή συνταγή. Και όπως είπε η Κάρμεν Φράγα, για τα επόμενα δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την Προεδρία του ICAT. Και αυτό δεν είναι ανέκδοτο. Είναι τα χρόνια 2014 και 2015 που θα συζητήσουμε θέματα πολύ σημαντικά, άρα λοιπόν αυτό το στοιχείο θα πρέπει να το κρατήσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μάουρο που ήρθε και που ετοίμασε την έκθεση. Αυτά. Merci. Euh, Ευχαριστώ, Ραούλ. Καταρχήν, σας ευχαριστούμε και τους τρεις που μας εκπροσωπούν. Είδαμε ότι είναι κάπως διαφορετικές οι απόψεις. Βέβαια δεν μας ε, εκπλήσει γιατί ο καθένας έχει την απόψή του. Βέβαια υπάρχει κάτι που με ανησυχεί γιατί εσείς ε, στα δίπλα-δίπλα στο αεροπλάνο της επιστροφής με τόσο αποκλείσεις απόψεις. Α, μάλιστα, όχι, όχι, κάνω. Αστιεύομαι, αστιεύομαι. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Μάλιστα, το γνωρίζω. Το αντίθετο. Και είστε οι δύο ειδικοί των θηνοειδών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και σας ευχαριστούμε. Ναι, ναι, ναι, το ίδιο σκεφτόμασταν. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Ο κύριος Άγνιου. Just before we break... Πριν διακόψουμε για φαγητό, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ το διερμηνέα που έκανε τη διερμηνία της κυρίας Φράγκα στα αγγλικά. Ήταν εξαιρετική η διερμηνία, διότι η κυρία Φράγκα μιλά πολύ γρήγορα και όποιος ήταν μπράβο του. 100%. Είναι αλήθεια ότι μιλάει πολύ γρήγορα η Κάρμεν. Κυρία Βράγκα, εγώ πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από του διαρμηνεί, γιατί ξέρω ότι δεν έχω αυτό έλεγχο όταν μιλάω. Μάλιστα, σα ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε το απόγευμα.